Colleagues, please be seated. Συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε. Παρά τη δυσκολία που είχαμε σήμερα με την αλλαγή των αιθουσών και την παρακολούθηση αλλεπάλληλων συνεδριάσεων, μας έχει μείνει ένα τελευταίο αλλά πολύ ενδιαφέρον σημείο στην ημερήσια διάταξη και ένα σημείο που μας ανησυχεί ιδιαίτερος. Με ιδιαίτερη χαρά λοιπόν έχω το προνόμιο να καλωσορίζω τον αντιστράτηγο Λούντβιχ Λάινχος που είναι επικεφαλής της υπηρεσίας ε, για τον κυβερνοχώρο και τις πληροφορίες των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων. Έχει μακρά πείρα ο στρατηγός. Είναι πολύ πύρο σε θέματα κυβερνοάμυνας. Μόλις είχαμε μια σύντομη συνομιλία και ελπίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να επεκταθούμε και πιο διεξοδικά σε θέματα κυβερνοασφάλειας. Για τα θέματα της κυβερνοασφάλειας και της κυβερνοάμυνας Περιλήθηκα και στην κοινή διακήρυξη του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν αναγνωριστεί ως α, ε, α, ε, σημαντική τομή συνεργασίας. Και θέλουμε να εξασφαλίσουμε κατάλληλο κοινοβουλευτικό έλεγχο αυτής της διαδικασίας. Παρόλο που κάποια πράγματα θα πρέπει να διευκρινιστούν και να διαλευκανθούν. Καλώς ήρθατε στρατηγέ μου και περιμένουμε πώς και πώς για να εκμεταλλευτούμε την πλούσια πείρα σας. Uh, Καλημέρα κύριε και κύριοι, είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι και πάλι στις Βρυξέλλες. Όπως θα γνωρίζετε κάποιοι, ήμουνα στο στρατηγείο του ΝΑΤΟ μέχρι το 2016 αυτό που θα κάνω σήμερα είναι να σας ε, παρουσιάσω τι έχουμε κάνει στη Γερμανία με μια προσέγγιση που περιλαμβάνει όλη την κυβέρνηση όσον αφορά την υπηρεσία μας. Θα ήθελα να ξεκινήσω με την ψηφιοποίηση. Είναι ένας όρος που αλλάζει το παιχνίδι στην κοινωνία μας. Και δεν είναι μόνο τεχνική πρόκληση, είναι μια πολύ ευρύτερη πρόκληση και αυτό δεν αφορά μόνο τους ε, πολίτες αλλά και το στρατό. Είναι μια τεχνική πρόκληση που θα έχει μεγάλο αντίκτυπο στην οργάνωση, στον οργανισμό μας, ε, στις διαδικασίες που ακολουθούμε. Επίσης θα πρέπει να συζητήσουμε και ποια είναι τα πιο πιθανά σενάρια και οι ε, σειράξεις που μπορούν να συμβούν μεταξύ ψηλά ψηφιμένων χωρών στο μέλλον. ποιε θα είναι οι συνέπειε τη ψηφιοποίησης. Θα έχουμε πολλά επαγγέλματα βέβαια που θα εξαφανιστούν ή που θα αλλάξει η φύση τους και που θα, πλήξουν προφανώς και του εργαζόμενου στο στρατό. Ε, ραγδαία είναι εξέλιξη τη ψηφιοποίηση στην κοινωνία μας. Λοιπόν, και αυτό φυσικά μας δίνει πολλά προνόμια αλλά έχουμε πάντα και τη δεύτερη πλευρά του νομίσματος, την αρνητική πλευρά του νομίσματος. Δεν θα ήθελα να σα δώσω όλα αυτά τα παραδείγματα. Έχω κάποιες διαφάνειες και μπορείτε να δείτε σε διεθνέ επίπεδο. Θα ήθελα όμως να σας δείξω το φάσμα των κυβερνοεπιθέσεων που μπορούν να συμβούν. Αυξάνονται και σε ποιότητα και σε ποιότητα. Και ξεκινάμε από κλοπή δεδομένων, χειραγώγηση πληροφοριών, άρνηση πρόσβασης, αλλά μπορεί να προκληθούν και κινητικά και ε, προβλήματα, εμπόδια και να θέσει, ε, να θέσει κανείς σε κίνδυνο και ζωές. Έχουμε παραδείγματα τέτοια. Είναι ευρύ το φάσμα λοιπόν. Και να δούμε το κομμάτι των πληροφοριών του κυβερνοχώρου. και έχουμε να αντιμετωπίσουμε και την επιρροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τα οποία ε, θέτουν σε τις δημοκρατικές μας αξίες στο πλαίσιο της ε, ραγδαίας ψηφιοποίησης. Υπάρχει μια ακόμα πρόκληση Έχουμε διάφορους παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν θέματα, από τα script και τους αριστέχνες hacker, το οργανωμένο έγκλημα, τους τρομοκράτες και τους κρατικούς ε, παράγοντες. Κάτι που πρέπει να γνωρίσουμε είναι ότι παράλληλα με το οργανωμένο έγκλημα και τα ε, κράτη και τους τρομοκράτες μπορούν να προκαλέσουν ε, ε, πολύ σοβαρά προβλήματα όλοι αυτοί οι φορείς στα υψηλά ψηφιοποιημένα κράτη, ειδικά και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας τώρα όσον αφορά τις ενοπλές δυνάμεις. Η ψηφιοποίηση δεν αφορά μόνο μία, έναν τομέα, αφορά όλη την κοινωνία, το κομμάτι της επικοινωνίας, τα συστήματα ελέγχου και βασικά θέματα του κλάδου, την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, τις υποδομές. Είναι ευρύ λοιπόν το φάσμα των δραστηριοτήτων πρέπει να λάβουμε υπόψη. Σε εθνικό επίπεδο Έχουμε δημιουργήσει ένα πλαίσιο στην πολιτική. Υπάρχει μια λευκή βουλή του 2016, μια εξαιρετική προσπάθεια και αν την ε, συγκρίνουμε με αυτή που είχαμε το 2006, μετά από 10 χρόνια λοιπόν που μεσολάβησαν, αν δούμε τον όρο υβριδικός ή cyber στην ε, Λευκή Βουλή 2006, ε, είναι όροι που δεν παρουσιάζονται καν. Ε, ενισχύει την προσέγγιση που εμπλέκει όλη την κυβέρνηση. και επίσης ε, ορίζει τι πρέπει να γίνει για να ενισχύσουμε τις δυνατότητες μας όσον αφορά επίσης και το προσωπικό. Δίνει και εκεί έμφαση σε αυτή την πρόκληση, κάτι που είναι πολύ σημαντικό και για την κοινωνία μας. Κάνει αναφορά στην αποδοτικότητα και ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε τους ε, πόρους μας για να το πετύχουμε αυτό. Υπάρχει ένα ακόμα έγγραφο το οποίο εκδόθηκε από το Κοινοβούλιο, Εθνικό Κοινοβούλιο του 2016, υπό την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Άμυνας. Και σε αυτό το έγγραφο, λοιπόν, υπάρχουν πολλά, ε, ε πολλές ενδιαφέρουσες ενολογικές προσεγγίσεις. Έχουμε πάλι και αυτή την προσέγγιση που συμπεριλαμβάνει όλη την κυβέρνηση, την περαιτέρω εξέλιξη ε, του Εθνικού Κέντρου Κυβερνοάμυνας σε στενή συνεργασία με τον Ομοσπονδιακό Στρατό, ε, ομάδες ε, αντιμετώπισης ε, περιστατικών. Επίσης, έχουμε λοιπόν ένα πορτφόλι που έχει να κάνει με όλα αυτά τα θέματα και το οποίο θα πρέπει να ερμηνευτεί και σε άλλους ε, τομείς. Είμαστε σε καλό δρόμο μέχρι στιγμής. Σε γενικές γραμμές βλέπουμε την ε, διακυβερνητική ευθύνη. Τρία υπουργεία αναλαμβάνουν την ευθύνη. Θα πρέπει βέβαια να υπάρξει κατάλληλο συντονισμός, το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο αντιμετωπίζει θέματα κυβερνοπολιτικής, κυβερνοασφάλειας είναι το Υπουργείο Εσωτερικών ε, υπεύθυνο γι' αυτό και έχουμε και για το θέμα της κυβερνοάμυνα, για το οποίο είναι υπεύθυνο το Υπουργείο Άμυνας. Είναι λίγο δύσκολο να διαφοροποιήσουμε μεταξύ άμυνας και ασφάλειας σε αυτό το τομέα. Έχουμε λοιπόν τη συνεργασία ε, αυτών των τριών φορέων, ε, που θα πρέπει να είναι σωστή για να έχουμε αποτελέσματα όσον αφορά την άμυνα. Το Υπουργείο Άμυνας αποφάσισε το 2015 να δημιουργήσει μια νέα ενέργεια για το πώς θα προσεγγίσουμε ως στρατός το θέμα αυτό και στις αρχές του 2018 ο υπουργό μας αποφάσισε ως ε, υπουργό μας πρώτα να δημιουργήσει μια διεύθυνση με έναν υπεύθυνο ε, πληροφοριών σε επίπεδο Υπουργείου Άμυνα και να δημιουργηθεί μια νέα στρατιωτική υπηρεσία στη Γερμανία για το κυβερνοχώρο και τις πληροφορίες. Όπως αποφασίστηκε και στις τελευταίες συνόδους του ΝΑΤΟ, Σύμφωνα με αυτή την απόφαση του ΝΑΤΟ, λοιπόν, κάναμε και εμεί, ε, ε, λάβαμε το κατάλληλο βήμα για να δημιουργήσουμε μια αντίστοιχη υπηρεσία Καταλαβαίνετε λοιπόν εδώ πέρα σε αυτή τη διαφάνεια ποια είναι η δομή στον Ομοσπονδικό Στρατό. Έχουμε το Υπουργείο, έχουμε τα ε, θέματα που αφορούν τον στρατό και αυτά που αφορούν τους πολίτες. Έχουμε τις δυνάμεις, έχουμε το στρατό, το ναυτικό, έχουμε την ε, ιατρική υπηρεσία, ένα κοινό κέντρο υποστήριξη θέματα διατομεακά και τελευταία έχουμε και την υπηρεσία κυβερνοχώρου και κυβερνοπληροφοριών. Είμαστε λοιπόν στο επίπεδο με τις υπόλοιπες υπηρεσίες ε, του στρατού και φυσικά έχουμε και άλλους ε, τομείς που είναι υπευθύνοι για το προσωπικό, για τις ε, προκηρύξεις και για άλλες δραστηριότητε. Σε αυτή την εικόνα θέλω να σας δείξω δύο πράγματα. Τον κυβερνοχώρο τον αντιμετωπίσουμε σαν έναν κλάδο όπως είναι ο αέρας, η γη, η θάλασσα, το διάστημα. Τι σημαίνει αυτό το ότι στον στρατιωτικό σχεδιασμό πάντα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη πώς θα χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες εκτός αυτών των τομέων. Είναι ένας ανεξάρτητος χώρος, ο οποίος όμως μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά ή συνοδευτικά στους κλασικούς τομείς ή να αντικαταστήσει ακόμα κάποιες δυνατότητες στους κλασικούς ε, τομείς του στρατού. Όσον αφορά τη δικιά μου την υπηρεσία, είναι μια μεγάλη οργάνωση ε, που λειτουργεί σε ταχύς ρυθμούς. Ξεκινήσαμε τον Σεπτέμβριο του 2015. Η απόφαση λήφθη τον Απρίλιο του 2016. Τον Απρίλιο του 2017 δημιουργήθηκε το επιτελείο και τον Ιούλιο ε, ανέλαβα εγώ. Uh, operational capability. Και θα ολοκληρωθεί ε, το έργο μας μέχρι το 2021. Είμαστε στη διαδικασία εργασιών, εξαρτώμαστε στην αρχή ε, από στήριξη από άλλες υπηρεσίες. Έχουμε φτάσει σε μια διάμεση κατάσταση που να προχωρήσουμε λίγο πιο γρήγορα και το 2021 πλέον θα έχουμε φτάσει ε, την ε, πλήρη επιχειρησική δυνατότητα. Ποιες είναι οι, οι ευθύνες της υπηρεσία μας. Υπάρχουν τέσσερις βασικοί πυλώνες. Η κεντρική αποστολή είναι να τρέξουμε το πληροφορικό σύστημα του Ομοσπονδιακού Στρατού, τις ε, υποδομές ε, πληροφόρησης του ε, στρατού και τις αφαιρές και τις κινητές. Επίσης, το θέμα της διασφάλισης του πληροφορικού μας τοπίου. Ένα δεύτερο, μια δεύτερη αποστολή είναι η διασύνδεση με τον κυβερνοχώρο τα μη κινητικά ε, But you can uh, reach... Το νέο, ο νέος που θα είναι ο χώρος της ε, κυβερνοασφάλειας. Έχουμε και ένα τρίτο πυλώνα της ε, γεωγραφικές ε, πληροφορίες, εντοπισμό θέσης, ε, βοηθάει το να έχουμε αντίληψη των καταστάσεων. Δεν παρέχονται μόνο γεωγραφικές πληροφορίες, αλλά και άλλες επιστημονικές, ε, επιστημονικοί κλάδοι καλύπτονται. Η υπηρεσία μας παίζει ρόλο στην κυβερνητική προσέγγιση για την ασφάλεια που σας έδειξα ότι διέπει τη θέση μας όπως ορίστηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών. Υπάρχουν διάφορες ε, δυνατότητες, ε, συλλογή πληροφοριών, ε, για ηλεκτρονικές επιχειρήσεις, ηλεκτρονικό πόλεμο, και διάφορες άλλες υπηρεσίες τις οποίες ε, τις συγκεντρώσαμε τώρα υπό την ομπρέλα, την ομπρέλα της δικής μας υπηρεσίας. Ποιες είναι οι δυνατότητες που αναπτύσσουμε περαιτέρω. Πέντε βασικοί τομείς. Ο πρώτος είναι να αναγνωρίσουμε καταστάσεις από την κρατική πλευρά. Θα επανέλθω σε αυτό. Για να δούμε τι επιχειρήσεις ενδεχομένω χρειάζεται να αναλάβουμε. Ενισχύουμε επίσης ε, το λογισμικό, όχι ε, ανταγωνιστικά προς τις βιομηχανίες, αλλά με εξατομικευμένες διαδικασίες προσαρμογής του λογισμικού στις ένοπλες δυνάμεις, ενίσχυση του πυλώνα κυβερνοασφάλειας, κάτι σημαντικό. Εκεί βάζουμε πολλές προσπάθειες. Επίσης, όπως είπα, και στην κλασική συλλογή πληροφοριών και σχέδες επιχειρήσεων εστιάζουμε. Αυτή είναι η βασική τομή που δραστηριοποιούμαστε. Τώρα θα ήθελα να μιλήσω λίγο για ε, την αναγνώριση της κατάστασης των τομέας και ασφάλειας. Ε, θα σας παρουσιάσω το τι κάνουμε με αυτή τη διαφάνεια. Υπάρχουν πολλοί τομείς που μπορεί να συνεισφέρουν ε, στην ευαισθητοποίηση για την κυβερνοασφάλεια. Μεταξύ των υπηρεσιών μας λοιπόν, στη δική μου υπηρεσία, έχουμε τα δικά μας συστήματα. Βλέπετε τα κέντρα για την κυβερνοασφάλεια. Έχουμε κέντρα πληροφοριών, υπηρεσίες πληροφοριών που μας δίνουν πληροφορίες σχετικά με τα, ό,τι αφορά τον κυβερνοχώρο και την κυβερνοασφάλεια. Θέλουμε να συγκεντρώσουμε αυτά τα στοιχεία ε, σε ένα κέντρο αντιμετώπιση ε, καταστάσεων, ένα κέντρο επιχειρήσεων και για καλύτερη ευαισθητοποίηση, αλλά και γιατί θέλουμε να παρέχουμε δείκτε προειδοποίηση αν κάτι συμβεί. Και βέβαια θέλουμε να υπάρχει συντονισμό ε, για τα αποτελέσματα που μπορεί να έχει μια δυνητική στρατιωτική επιχείρηση κτλ. Βέβαια, βλέπουμε τη στρατιωτική εικόνα, αλλά την εντάσσουμε σε μια πιο ολιστική προσέγγιση. Και όλα αυτά ε, τα εκπεξεργάζεται το κέντρο ε, καταστάσεων στο ΣΥΝΤ που υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Έχουμε τώρα διάφορους ε, πελάτες και στις ένοπλες δυνάμεις ε, και εκτός ε, των ομοσπονδιακών ενόπλων δυνάμεων. Μια άλλη πτυχή που θέλω να αναφέρω είναι το προσωπικό. Έχουμε προκλήσει σε πολλούς τομείς. Είναι μεγάλες οι απαιτήσει για εμπειρία και τεχνογνωσία. Ιδίω για τη συγκρότηση των δυνάμεων. Και ένας από τους λόγους για τους οποίους έχουμε τη δική μας υπηρεσία είναι γιατί στο γερμανικό σύστημα μπορείς να ασκήσεις επιρροή και να αλλάξεις ε, επαγγελματικές σταδιοδρομίες μόνο αν είσαι ε, αρχηγός επιτελείου και έχεις ένα ρόλο σε αυτό. Θέλουμε λοιπόν να αλλάξουμε την ε, σταδιοδρομία και το μονοπάτι της σταδιοδρομίας στο στρατό και φυσικά μας δίνουν οι μη στρατιωτικοί συνάδελφοι την πολύτιμη εμπειρία τους στο σχεδιασμό προσόντων και της εκπαίδευσης και ζητούμε επίσης ε, κίνητρα, παρακολουθούμε τα κίνητρα, έχουμε δραστηριότητες εκπαιδευτικέ και άλλες ε, για να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον. Πολλά γίνονται, άλλα έχουν ξεκινήσει εν μέρη, άλλα είναι ακόμα στα σκαριά. Μια συγκεκριμένη πτυχή θέλω να αναφέρω, την αρχή του 2018 στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου έχουμε ένα μάστερ για την, ένα μεταπτυχιακό για την κυβερνοασφάλεια, όχι μόνο για στρατιωτικούς, αλλά και για κυβερνητικούς κρατικούς οργανισμούς, για ευαισθητοποίηση στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Και ελπίζουμε βέβαια να αποφυτίσουν και να πάρουν το μεταπτυχιακό τους ε, όσοι φοιτούν σε αυτό το πρόγραμμα. Είναι μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση και με μεγάλη αποδοχή για Ένα άλλο τομέα είναι κυβερνο... κυβερνότητα του κυβερνοχώρου, η Cyber Reserve. Πάντα ε, σε αυτή την ε, προσέγγιση που ελαμβάνει όλη την κυβέρνηση θέλουμε ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών. Έχουμε μια κοινότητα εμπειρογνωμόνων. Δεν μας ενδιαφέρουν όμως ε, μόνο οι στρατιωτικοί, αλλά και το προσωπικό που εργάζεται στο μη στρατιωτικό τομέα, αλλά έχει αποκτήσει τεχνογνωσία και εμπειρία ως πολίτης. Μας ενδιαφέρουν και άλλοι που δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία και θέλουμε να τους εντάξουμε στο σύστημα. Είναι μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Από τότε που ιδρύθηκε η υπηρεσία μας είχαμε πάνω από 500 αιτήσει, μόνο και μόνο γι' αυτό. Το θέμα και πάνω από 100 άτομα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο συμμετέχουν στο σύστημα. Cyber cluster, ο κυβερνομάδα είναι κάτι άλλο στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου. Μίλησα για το μεταπτυχιακό και στην κυβερνοασφάλεια. Υπάρχει όμως και κάτι ακόμη. Μια πλατφόρμα στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου που εκεί θα συναντά η βιομηχανία, την επαγγελματική κοινότητα και το εκπαιδευτικό σύστημα πανεπιστημίου των ελληνικών Δυνάμεων για να έχουμε μια καλύτερη διαδικτύωση και μια τέτοια προσέγγιση. Να εκμεταλλευτεί δηλαδή ο ένας τις εμπειρίες του άλλου. Εκπαίδευση, κατάρτιση, επιστήμη. Εκεί εστιάζουμε. Αλλά έχουμε μια εγκάρσια τοποθέτηση στο Μόναχο. Ένας άλλος τομέας είναι η καινοτομία στον κυβερνοχώρο και έχουμε το σχετικό κόμβο στι ομοσπονδιακές άνοπλες δυνάμεις. Είναι μια δραστηριότητα που λειτουργεί πιλωτικά τα τελευταία τρία χρόνια για να έχουν οι ένοπλες δυνάμεις την εμπειρία μιας νεοφυούς επιχείρησης για να βελτιώσουμε την καινοτομία, κάτι που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για τους δικούς μας σκοπούς. Και θέλουμε να εντάξουμε αυτό, αυτούς τους ανθρώπους και στις κοινότητες του κυβερνοχώρου γιατί είναι άνθρωποι με πολλά ταλέντα και δεξιότητες που μπορούν να βοηθήσουν. Τρία χρόνια λοιπόν είναι η αρχική φάση, η πιλωτική και θα δούμε πώς θα συνεχίσουμε μετά. Θα εξαρτηθεί από το πώς θα, ποια θα είναι η έκβαση αυτού του προγράμματος. Ίσως έχουμε ένα ειδικό τμήμα μετά. Διεθνή συνεργασία. Ήδη ξεκινήσαμε τη συνεργασία μας με τους εταίρους μας από τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση διάφορες μορφές συνεργασίας. Χθες, για παράδειγμα, γύρισα από το Ταλίν, που εκεί είδα τις διοικήσεις κυβερνοχώρων από τις χώρες των ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες χώρες. Χθες πήρα τη σκητάλη εγώ στη θέση του Προέδρου μετά την Ολλανδία. Κάθε χρόνο αλλάζει η Προεδρία. Άρα εμείς θα είμαστε Προέδρη, Η Γερμανία θα προεδρεύει αυτού του φόρουμ των διοικητών του κυβερνοχώρου. Στηρίζουμε επίσης και από τις πιο μικρές χώρες. Δηλαδή στη δημιουργία υποδομών, capacity building λέμε, μπορεί και εσείς να χρησιμοποιείτε αυτό το όρο στην Ένωση. Λίγο πολύ αυτή είναι η ολιστική προσέγγιση που ακολουθούμε ε, μάλλον συνεργάζομαι και με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Έχουμε ανταλλαγή με διάφορου ε, άλλου ε, φορεί. Νομίζω ότι είναι μια υποχρεωτική προσέγγιση, απαραίτητη προσέγγιση, να μην προσπαθούμε απλά να ευαισθητοποιήσουμε γενικώ την κοινωνία, αλλά και να αντιμετωπίσουμε τα κοινά συμφέροντα. Αυτά ως ε, παρουσίαση. Φυσικά είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω στις απορίες σας και να συμπληρώσω αυτή την παρουσίαση. Ευχαριστώ. Wow. Ε, δεν έχουμε και μεγάλη επιλογή. Φαντάζομαι ο κύριος Γκάλερ θα θέλει να μιλήσει Ευχαριστώ πολύ για την ενδιαφέρουσα παρουσίαση. και την πληροφόρηση για το πώς αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση στη Γερμανία και επίσης ε, στο γεγονός ότι θα χρειαστούν πολλές συνεργασίες στον ε, τομέα. Επιστρέψτε από την Ιταλία. Υπάρχουν, ε, υπάρχει στήριξη και από άλλες χώρες για την δημιουργία των κατάλληλων υποδομών. και κάποιε άλλε μπορούν να παρέχουν περισσότερη αναπτυξιακή βοήθεια γιατί είναι πιο ε, ανεπτυγμένοι στον τομέα αυτό. Προκύπτουν κάποια ερωτήματα. Ένα αφορά τη συνεργασία κατά πρώτον, πώ θα μπορούμε να το πετύχουμε και να το οργανώσουμε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. όπω είναι αυτά τα φόρμ στα οποία προεδρεύεται. Πώς θα μπορούμε να τα διευρύνουμε αυτά σε άλλες ε, περιφέρειες, σε άλλους τομείς της ζωής, ε, του δημόσιου είναι δύσκολο να δημιουργήσουμε κάποιους περιορισμούς, κάποια όρια, ποιος συνεργαστεί με ποιον κτλ. Υπάρχει κάποια αρχή την οποία έχετε αναπτύξει ε, σύμφωνα με την οποία θα οριοθετήσετε ε, το ποιος θα συμβάλλει σε αυτή την ε, συνεργασία. Επίσης θα με ενδιέφερε να μάθω από πότε θα ξεκινήσουμε να συζητούμε για το θέμα. Αν συμβεί τους χάρη μια τεράστια κυβερνοεπίθεση, επίθεση, η παραβίαση του άρθρου 5, ε, μπορεί να συγκριθεί με μια τέτοιου είδους παραβίαση. Νομίζω ότι δεν υπάρχει συμφωνία σε αυτό το θέμα. Μπορείτε να μου πείτε σε ποια κατεύθυνση θα οδηγηθεί η συζήτηση σε περίπτωση μιας επίθεσης. Και επίση, ε, ως προς το πρακτικό κομμάτι, υπάρχουν παραδείγματα ε, από φέτος ε, που δέχτηκε επιθέσεις, ε, γεωνοπιθέσεις η Γερμανία από τη Ρωσία. αν κάποιος ανακαλύψει ότι έχει συμβεί κάτι τέτοιο, εσείς είστε ο πρώτος που θα πληροφορηθεί. Δεν ξέρω ποια είναι η των πληροφοριών, δηλαδή από πού προς τα πού ρέουν οι πληροφορίες σε περίπτωση τέτοιων περιστατικών. Για τέτοιου είδους ε, ε, επιθέσεις δεν αφορούν μονάχα μία χώρα. Αν υπάρχει συνεργασία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ΝΑΤΟ. Επειδή είναι ένα πολύ ευρύ φάσμα το οποίο καλύπτει αυτή η πρόκληση, επανέρχομαι και πάλι στο ερώτημα πώς οριοθετούμε τις δραστηριότητες ώστε να υπάρξει αποτελεσματική ε, αντιμετώπιση της κατάστασης. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Δρογεύσκη. Με συγχωρείτε. Τα γερμανικά μου δεν είναι τόσο καλά. Γι' αυτό θα μιλήσω στα πολωνικά. Με συγχωρείτε. Η πρώτη μου ερώτηση αφορά ε, έναν έπαινο που θέλω να σας κάνω πολύ καλή και μεθοδική απάντησή σας, ε, η γερμανική απάντηση στις κυβερνοαπειλές. Πολύ καλός ε, καταμερισμός αρμοδιοτήτων, καλή κατάρτιση εκπαίδευση, ε, με έφθετο χρονοδιάγραμμα. Πολύ καλό το έγγραφο. Θα μπορούσε να γίνει δεκτό και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μπράβο σας λοιπόν. Πάντως αυτό το περίπλοκο σύστημα θα μπορούσε να μεταλαμπαδευτεί και σε άλλες χώρες γιατί ή μήπω ανταποκρίνεται σε ε, γερμανικές ιδιαιτερότητες. Μπορεί να γίνει ένα μοντέλο και για τους υπόλοιπους. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Δεύτερον, στην προηγούμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας λάβαμε την πληροφορία ότι κάποιες ε, τρομοκρατικές οργανώσεις ε, ξοδεύουν ε, δεκαπλάσια χρήματα για την παρουσία τους στο διαδίκτυο. Με στρατολόγηση, με προπαγάνδα από ό,τι ασχολούνται με ε, τρομοκρατικές επιθέσεις. Αυτή τη στιγμή ε, οι αναλογίες ε, πώς έχουν σε σχέση με τις προοπτικές για τα επόμενα 3-4 χρόνια. Ποιες είναι οι προβλέψεις που κάνετε για τη Γερμανία. Υπάρχει αύξηση των δαπανών στην κυβερνοασφάλεια. Τρίτη ερώτηση. Ε, μια σημαντική διάγνωση. Όσο επεκτείνεται η παγκοσμιοποίηση, όσο έχουμε πρόσβαση σε συγκεκριμένα προγράμματα, τόσο πιο δύσκολο θα εξασφαλίσουμε την ασφάλειά τους. Από άποψη άμυνα και ασφάλειας, με τη διασταλτική ευρεία έννοια. Σήμερα θα πρέπει να απομακρυνθούμε από την παγκοσμιοποίηση για να θωρακιστούμε απέναντι σε ε, κυβερνοεπιθέσεις, ε, κυβερνοαπειλές ε, και από και τα, τα κυβερνητικά συστήματα, τα οικονομικά συστήματα, καλύτερη επιτήρηση. Πρέπει να απομακρυνθούμε από την ε, παγκοσμιοποίηση. Επίσης, ό,τι αφορά τα δορυφορικά συστήματα, ξέρω ότι η, ο γερμανικός στρατός στηρίζεται στο GPS, δηλαδή στο δορυφορικό σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών. σε ποιο βαθμό η επιτυχία του Κοπέρνικος και του Γαλιλαίου θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από το γερμανικό στρατό, από το γερμανικό κράτος και από την Ευρώπη για να αντιμετωπιστούν οι απειλές και όχι μόνο οι τρομοκρατικές απειλές. Σας ευχαριστώ κύριε Στρογεύσκη. Δεν έχουμε άλλα μέλη στην αίθουσα, οπότε δεν έχουμε άλλες ερωτήσεις από την ομίγυρη. Θα κάνω και εγώ κάποιες ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ στρατηγέ μου για την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ενημέρωση που μας κάνατε. Και θα ήθελα, δεδομένη της πλούσιας εμπειρίας που έχετε, να μας πείτε ποια είναι η γνώμη σας για τα προβλήματα που έχουμε και τις δυσκολίες ό,τι αφορά την αντιμετώπιση επιθέσεων. Και ότι μερικοί ιδιοποιούνται ή αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις κυβερνοεπιθέσεις ε, και σε σχέση με αυτά που είπε και ο κύριος Σδρογεύσκη για τη συμμετοχή κάποιων ε, κρατικών φορέων ή κυβερνητικών φορέων. Και έχουμε από τη μια την κυβερνοασφάλεια και την κυβερνοάμυνα. Πείτε μας ε, δύο λόγια και γι' αυτό. Την αντιπαραβολή κυβερνοασφάλειας και κυβερνοάμυνας. Ε, το πρωί μιλήσαμε για τις συνέπειες του Brexit στην κοινή, ασφάλεια, ε, στην κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Εσείς ε, πιστεύετε ότι μετά το Brexit θα αλλάξει το modus operandi στα θέματα αυτά, της κυβερνοασφάλειας δηλαδή, αλλά και της ανταλλαγής πληροφοριών των μυστικών υπηρεσιών. και σε τι επίπεδο θα γίνεται, σε επίπεδο συνεργασίας ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιο κατά τη γνώμη σας είναι το κατάλληλο επίπεδο συνεργασίας για να αντιμετωπίσουμε τις σοβαρές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Αυτά προς το παρόν και σας ακολουθήσει και δεύτερος γύρος ερωτήσεων. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Θα περάσω στα γερμανικά τώρα, αν μου επιτρέπετε. Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα για την οριοθέτηση και για το ποιος θα συμμετέχει στις ε, ενέργειες, θα υπάρξει μια διαφοροποίηση στη φάση που ακόμα δεν έχουν βρεθεί λύσεις. Θα πρέπει να ε, καθιερώσουμε στην αρχή έναν διάλογο και μετά να συνεχίσουμε με την οριοθέτηση. Γιατί αυτά τα θεματικά παιδεία δεν ε, εντάσσονται στο comfort zone αυτό που πρέπει να λάβουν τις αποφάσεις. Πιο συγκεκριμένα... Για τους μηχανισμούς, αυτό που έχουμε στη μέχρι στιγμής, έχουμε ένα εθνικό κέντρο στο οποίο είναι παρόντες όλοι οι θεσμοί που ασχολούνται με την άμυνα, η εγκληματολογική υπηρεσία κτλ. Και αυτός είναι ο μηχανισμός μας για να ενορχιστρώσουμε και να συντονίσουμε τέτοια θέματα. Όσον αφορά το άρθρο 5 για τις κυβερνοεπιθέσεις, στο ζήτησαμε όταν ήμουν εδώ πριν από κάποια χρόνια, είναι απόφαση Υπουργών Κυβερνήσεων. Υπάρχει ένα ανοιχτό ερώτημα για το ποιο είναι το κατόφλητο όριο. Γιατί δημιουργείται κάποιο ρίσκο όσον αφορά μια ενδεχόμενη κυβερνοεπίθεση και θα πρέπει φυσικά να υπάρχει ένας βαθμός δυσκολίας και είναι μια ουσιαστικά αποτρεπτική προσπάθεια ε, επίδραση αυτή που έχει, αλλά θα πρέπει να ορίσουμε ποιος θα αντιδράσει σε αυτό και γι' αυτό δεν υπάρχει ένας ακριβής ορισμός ως προς το ποιος θα αντιδράσει σε περίπτωση κυβερνοεπίθεσης. Τώρα σαν αφορά την ερώτηση του Πολουνού συναδέλφου, ευχαριστώ για το κομπλιμέντο. Όσον αφορά τι άλλε χώρε, είναι ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει εκεί και αν η συνάντηση με του συναδελφού μου από τι άλλε χώρε. Ε, Πώ θα πάει. Υπάρχει το θέμα το οργανωτικό το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε στη Γερμανία, αλλά θέλουμε να δούμε και πώς θα λειτουργούν τα υπόλοιπα κράτη, να δούμε ένας προς έναν τι ε, πράττουν στον τομέα. Π.χ. η Αμερική, η οποία είναι ήδη ενεργή σε αυτόν τον τομέα, να δούμε πόσο γρήγορα μπορεί να εφαρμοστούν όλα αυτά. Είναι δύσκολο να το προσδιορίσουμε ακόμα, γιατί η πρόκληση μεγάλη όταν έχουμε ε, μια μεγάλη οργάνωση, η προσέγγιση είναι από τα πάνω προς τα κάτω, είναι top-down προσέγγιση. Είναι θέμα επίσης διοίκησης, πολιτικής διοίκησης στις εκάστοτε χώρες, πώς θα δημιουργηθεί η αντίστοιχη δομή. Αλλά προφανώς θα ε, γίνεται σύγκριση ένας προς έναν και να δούμε πώς ε, θα προσεγγίσουμε και το θέμα της ε, στρατιωτικής διοίκησης. Θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Δεν ξέρω αν είμαστε σωστοί 100% ως προς ε, τον τρόπο που ακολουθούμε, αλλά θεωρούμε ότι μέχρι στιγμής προχωράμε καλά όσον αφορά τα κέρδη από την τρομοκρατία και το ίντερνετ. Δεν μπορώ να την απαντήσω γιατί είναι μια ερώτηση που έχει να κάνει με τις υπηρεσίε πληροφοριών και είναι δύσκολο να μιλήσουμε γι' αυτό σε μια ανοιχτή συνεδρίαση. Παγκοσμιοποίηση. Και η παγκοσμιοποίηση αποτελεί μια πρόκληση. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε την παγκοσμιοποίηση. Όμως έχουμε πολλές πλευρές που πρέπει να δούμε διαφορετικά. Έχουμε αναπτύξει συστήματα και στον αστυνομικό τομέα όσον αφορά την ασφάλεια. Αν και δεν ήμασταν αρκετά προχωρημένοι στο συγκεκριμένο κλάδο ως ε, στρατός. Τώρα όμως που έχουμε βρεθεί στο επίκεντρο του ανταγωνισμού, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι και στον κλάδο της κυβερνοασφάλειας Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι ένα παράγοντα επιβίωση και για τη βιομηχανία και για άλλου τομεί κλάδου τη οικονομία. γιατί υπάρχει ο κίνδυνος και υπάρχει περίπτωση να υπάρξουν ε, οικονομικές απώλειες. Γι' αυτό είναι σημαντικό να μην σταματήσουμε την παγκοσμιοποίηση αλλά να δημιουργήσουμε μηχανισμούς διασφάλισης ε, πρότυπα ώστε να περιορίσουμε τον ε, κίνδυνο. Υπάρχει ένα υπόλοιπο ποσοστό κινδύνου, θα πρέπει όμως να το περιορίσουμε όσο γίνεται. Πάντα πρέπει να προκύπτουν καινούργιοι μηχανισμοί. Όπω και στο σπίτι μας πρέπει να επικαιροποιούμε, να κάνουμε update στο αντιβάρου στο σύστημα. Παρ' όλα αυτά, το θέμα της κυβερνοσφάλειας είναι ένας θεμέλιος λίθος που είναι πολύ σημαντικό σε εθνικό επίπεδο σαν αφορά τον Γαλιλαίο. Είναι ένα θέμα στο οποίο θα πρέπει να προχωρήσουμε. Μία ακόμα ερώτηση. τα ερώτηση που έχουμε στον τομέα είναι το θέμα της ταχύτητας σε περίπτωση επιθέσεων, αν ξέρουμε όλες τις, ε, τις προϋποθέσεις για να ξέρουμε ποιος είναι αρμόδιος για τη διαχείριση του θέματος. Είμαστε οργανωμένοι ως κράτος ώστε να υπάρχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες όταν γνωρίζουμε τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις και τους συγκεκριμένους όρους. Όταν δεν γνωρίζουμε τους όρους, πάλι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις καταστάσεις και αυτό είναι μια πρόκληση που έχουν να αντιμετωπίσουν τα κράτη όσον αφορά το θέμα του attribution, και το, δεν, είναι, δεν είναι σαφής και επίσης υπάρχει το θέμα των συνόρων που δεν είναι σαφή, τότε υπάρχει ακόμη περισσότερο πρόβλημα στην, ε, στον ορισμό, στο να προσθέσουμε τις αρμοδιότητες. Όσον αφορά τους ε, παράγοντες, έχουμε και εκεί προβλήματα με κλασικέ ε, στρατιωτικέ επιθέσεις εδώ και δεκαετίε. εκατονταετίες και τώρα έχουμε μια νέα πρόκληση όπου μη κρατικοί φορείς έχουν πιο απλά μέσα στη διάθεσή τους ε, για να επιτεθούν. Επίσης μια πολύ σημαντική πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, το Brexit. Θα μπούμε σε πολιτική συζήτηση είναι μέλο του ΝΑΤΟ του Ηνωμένο Βασίλειο. Θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε κανονικά από συνδική πλευρά. Υπάρχουν και φυσικά και διμερεί σχέσει που υπάρχουν με το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν έχουμε επομένω ε, αρνητική συνέπεια από τον Brexit στο στρατιωτικό τομέα. Τα υπόλοιπα πολιτικά θέματα είναι πιο πολύ δικό σα ε, θεματικό πεδίο. Okay. Our colleagues... Καλώς. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις προς το καλεσμένο μας. Ο κύριος Γκάλερ. Ένα άλλο θέμα που αναφέρατε αυτό το cyber reserve, η κοινότητα του κυβέρνου χώρου, μιλάμε για αυτούς ε, τους εφέδρους. Ε, είναι ένας τομέας κλασικός ε, μπορεί να μην έχει να κάνει ακριβώς με τις ένοπλες δυνάμεις, αλλά υπάρχουν κάποιοι που είναι οι δήμονες σε αυτό το τομέα, είναι ειδικοί. Ε, επομένως, συγκεκριμένα εφέδρους θα μπορούσε να τους χρησιμοποιήσει στον τομέα αυτό ή γενικώ στον τομέα της βιομηχανίας, της μη στρατιωτικής ε, θα μπορούσατε να προσανατολιστείτε και με βάση τις ε, τελευταίες εξελίξεις για να είναι ενήμεροι η πρόεδρος. Ναι, μπορείτε να απαντήσετε. Είναι ένα ευρύ φάσμα. Έχουμε τους ε, κλασικούς εφέδρους ε, που έρχονται, αλλά υπάρχουν και κάποιοι που είχαν κάνει κάτι τελείως διαφορετικό ε, όταν ήταν σε ένοπλες δυνάμεις ε, και μετά κάνουν κάτι τελείως διαφορετικό. Δεν θέλουμε κλασικούς εφέδρους. Υπάρχουν και κάποιοι που δεν ήταν σε ένοπλες δυνάμεις, αλλά τους ενδιαφέρει το ζήτημα αυτό. Ε, και θέλουν να συνεισφέρουν στις ενόπλες δυνάμεις και υπάρχουν διαφορετικοί μηχανισμοί ε, για το πώς μπορούν ε, να αξιοποιηθούν μέσω συμβάσεων και τα λοιπά οι δεξιότητές τους. Και κάθε φορά βλέπουμε κατά περίπτωση το ζήτημα και Έχουμε αυτούς τους 500 ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονταν, αλλά είναι αρκετά κουραστικό και παίρνει χρόνο να εξετάσουμε την κάθε περίπτωση. Για τους κλασικού αφαίρου είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Αλλά υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις που πρέπει να καλυφθούν κάποιοι τομείς ε, λοιπά Υπάρχουν ε, κάποιες απαιτήσει. Αλλά προσπαθούμε ε, με τους συγκεκριμένους εμπειρογνώμονες να έχουμε κάποια ειδική μορφή σύμβασης και συνεργασίας. Επίσης έχουμε πολλές επαφές με εταιρείε ειδικέ. Σίγουρα το θέμα της συμμόρφωσης μας ενδιαφέρει και εξετάζουμε και δομής Τομεί, μάλλον που μπορεί να μην έχουμε εμεί κάποια συμβασιστική σχέση, αλλά έχουν κάποια εμπειρία, όπω οι τράπεζες για παράδειγμα. I think there are no... Δεν νομίζω να υπάρχουν, λέει άλλοι που να ζητούν το λόγο, γελώντα το λέει εκ μέρου τη Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πραγματικά θερμά στρατηγέ για τη γενική αυτή επισκόπηση και παρουσίαση της εκτεταμένης εμπειρίας σας και της ε, αλλαγής αυτής ε, πνεύματος ε, στις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον που προσπαθούμε να ε, μιμηθούμε κι εμείς, ε, υπάρχει μεγάλη εστίαση στο θέμα της ε, ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και προσπαθούμε όλοι να συλλέξουμε εμπειρίες σε επίπεδο ένωσης και από το ΝΑΤΟ και να τις αξιοποιήσουμε τις εμπειρίες αυτές και στις δικές μας συζητήσεις και αποφάσεις. Υπάρχει βελτιωμένη συνεργασία, ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά προσπαθούμε επίσης και να καταγράψουμε την εμπειρία των κρατών μελών και να την αξιοποιήσουμε. Ευχαριστώ για μια ακόμη φορά λοιπόν. Αγαπητοί συνάδελφοι, υπό τα διάφορα υπάρχει κάτι. Όχι. Επόμενη συνεδρίαση. Α, κάτι λέει ο Γραμματέας. Τρίτη, 15 Μαΐου. Σας περιμένουμε όλους. Ευχαριστώ τους Δερμηνείς, ευχαριστώ και τη Γραμματεία για τη σκληρή δουλειά. Πέρα τη συνεδρίαση.